Let uh, Σας ευχαριστώ. Ε, ξεκινάμε τη συνεδρίαση της ε, Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και της ειδική Επιτροπής για την ε, Φοροαποφυγή και Φοροδιαφυγή, της οποίας θα προεδρεύσουμε δύο Τσέχοι, ο κύριος Γέτσεκ και εγώ. Να σας πω ότι έχουμε 11 γλώσσες διαθέσιμες. Η συνεδρίαση αναμεταδίδεται στο ε, site του Ευρωκοινοβουλίου και επίσης θα έχουμε και ε, τα πρακτικά της συνεδρίασης στα αγγλικά. Θα δώσω το λόγο στον Πίτρα για να εξηγήσει για ποιο λόγο διοργανώσαμε τη σημερινή κοινή ακρόαση. Σας ευχαριστώ. Να σας καλωσορίσω όλους στην κοινή ακρόαση της ΕΚΟΝ και της ΤΑΞ 3. Θα συζητήσουμε το σκάνδαλο Κουμέξ, ε, οικονομικό έγκλημα και παραθυράκια στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ο στόχος αυτής της ακρόασης είναι να εξετάσουμε τις πρόσφατες αποκαλύψεις για τους φακέλους Κουμέξ που έδειξαν ότι πάνω από 55 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν πέσει αντικείμενο απάτης μέσω διαφόρων ε, ε, σχεδίων. Αυτή η ακρόαση στόχο θα έχει να εξετάσει τις υφιστάμενες νομικές ε, ευκαιρίες που επιτρέπουν τέτοιες, τέτοιου είδους καταστάσεις η ακρόαση θα αποτελείται από μόνο ένα πάνελ που αποτελείται από τρεις εμπειρογνώμονες. Ο πρώτος είναι ο κύριος Γκέρχαρτ Σίκ που είναι μέλος της Γερμανικής Βουλής, μέλος και συνεισηγητής της ε, πρώην Επιτροπής Έρευνας του Γερμανικού Κοινοβουλίου για το σκάνδαλο Κουμέξ. Παρόν εδώ είναι ο κύριος Χρήστοφ Σπέγγελ, που είναι ερευνητής στο ZW και πρόεδρος της έδρας Business Administration και Φορολογία 2 στο Πανεπιστήμιο του Μανχάιμ και ο κύριος Όλιβερ Σρέμ που είναι ιδρυτής και επικεφαλής της Διεθνούς Συνεργασίας του Project Cumex, Cumex καθώς και επικεφαλής συντάκτης του ε, δημοσιογραφικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού της Γερμανίας που ονομάζεται Corrective. Επίσης συνοδεύεται από τον κύριο Κρίσιαν Σαλεύσκη που είναι δημοσιογράφος και ρεπόρτερ στο Πανόραμα και στο Insight και είναι επίσης ε, τμήμα ε, του, των φακελών Κουμέξ. Ο κάθε ομιλητής θα έχει maximum 7 λεπτά για την εισήγησή του. και μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση. Θα πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Σικ θα είναι διαθέσιμος μέχρι τις 8. Οπότε οι συνάδελφοι που θα ήθελαν να του υποβάλουν ερωτήσεις θα πρέπει να το πράξουν μέχρι εκείνη την ώρα. Τώρα λοιπόν θα δώσω το λόγο στον κύριο Σίκ για την ε, επτάλεπτη εισήγησή του. Παρακαλώ. Αγαπητέ Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτέ, σα ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σα την εμπειρία μου σε σχέση με το, κουμ, το σκάνδαλο Κουμέξ και Κουμκουμ, σκάνδαλο που μα κόστησε εμά, του φορολογούμενου, δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν ξεκίνησα την κοινοβουλευτική έρευνα για τα Κουμέξ στη Γερμανική Βουλή, το κίνητρό μου δεν ήταν να ανακαλύψω εγκληματικέ δραστηριότητε του παρελθόντο. Αυτό θα πρέπει να το κάνουν οι εισαγγελεί και το το, ο εισαγγελέα της κολονίας κάνει εξαιρετική δουλειά κατά την άποψή μου. Η πρόθεσή μου ήταν να με εξασφαλίσω ότι θα μάθουμε από τις ε, αποτυχίε των δημοσίων θεσμών και να ε, προλάβουμε παρόμοιες υποθέσεις στο μέλλον. Η ιστορία των ε, μερισμάτων ε, στη Γερμανία από τις αρχές του 90, τις δεκαετίες του 90 μας δείχνει ότι οι διάφοροι dealer έχουν ε, μεταβάλει τις προσεγγίσεις τους προσαρμοζόμενοι ομαλά στις αλλαγές στην νομοθεσία και στους διοικητικούς μηχανισμούς. Θα ήταν αγαθό να υποθέσει κανείς ότι η νομοθεσία που σταμάτησε το cum στη Γερμανία το 2011 και ο νόμος ο οποίος προσπάθησε να περιορίσει τα κουμ το 2016 θα μπορούν μάλλον να εμποδίσουν τέτοιες δραστηριότητε στο μέλλον. Από τη στιγμή που οι εποπτικές αρχές και οι υπεύθυνοι των φορολογικών γραφείων ε, δεν ε, με την ίδια ταχύτητα, δεν θα μπορέσουν να κερδίσουν τον αγώνα ενάντια στους εμπειρογνώμονες ε, Τη οικονομία, οι οποίοι διαρκώ σχεδιάζουν νέα τρίκ για να γεμίζουν τι τσέπε τους και να βριάζουν τι τσέπε των φορολογούμενων δεν με εξέπληξε λοιπόν καθόλου όταν ένα νέο μηχανισμός αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα. Ένα τρίκ που πάλι, ε, όχι προς έκπληξή μας, ξεκίνησε περίπου τη στιγμή που σταμάτησαν το cum το 2011. Αυτή τη φορά το τρίκ είναι να δημιουργηθούν ε, παραπάνω από μία αποδείξη ε, απόθεσης μερισμάτων ανά μέρισμα, ανά Το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας κατάλαβε αυτό το θέμα μέσω, αυτή την απάτη μάλλον, μέσω των ε, δημοσιογράφων έρευνας και όχι μέσω κάποιου ελεγκτή. Το Υπουργείο Οικονομίας πίστευε πως ε, είχε κάνει τη δουλειά του όταν σταμάτησε τα ΚΟΜΕΚ το 2011. Τα πορίσματα της ε, Κοινοβουλευτικής Ερευνητικής Επιτροπής αγνοήθηκαν, ακόμα και αν είχαν ε, προκύψει πολλά μειονεκτήματα και προβλήματα. Θα σας αναφέρω κάποια απορίσματα που μπορεί να σας, σας χρησιμεύσουν. Καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Συνεργασία. Το 2005 οι Ολλανδικές εφημερίδες έγραψαν για μια απόφαση δικαστηρίου για την απόλυση ενός τραπεζικού υπαλλήλου. Οι δημοσιεύσεις έδειξαν ότι στη διάρκεια της υπόθεσης το εμπόριο κουμέξ έπαιξε ρόλο. Εάν οι γερμανικές αρχές είχαν ακούσει αυτή την υπόθεση θα είχαν αντιδράσει πολύ νωρίτερα. Το 2008 η Ελβετία σταμάτησε τα κουμέξ και έτσι προστάτευσε τους, τους Ελβετούς φορολογούμενους. Η Γερμανία αγνόησε αυτή την κίνηση και τις πήρε ακόμα τρία ε, πολύ δαπανηρά χρόνια μέχρι να σταματήσουν αυτού του είδους το εμπόριο στη Γερμανία ε, εμπόριο το οποίο εν μέρη οργανωνόταν από τις ελβετικές τράπεζες. Οι δανείοι φορολογούμενοι έχασαν 1,7 δις ευρώ όταν οι ίδιοι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στη Γερμανία μέχρι το 2011 μετακινήθηκαν προς εκεί. Η ευρωπαϊκή συνεργασία λοιπόν θα είχε σώσει, θα είχε γλιτώσει τους Ευρωπαίους φορολογούμενους από πολλά, ε, ε, ε πολλές τέτοιες ζημιές. Η ηγεσία του Μπάφιν, δε, της Γερμαν... του Γερμανικής Εποπτικής Αρχής, δεν είχε ιδέα τι συνέβαινε. Ακόμα και όταν οι εφημερίδες ανέφεραν τι γινόταν με τα Κουμέξ, θεώρησαν ότι ήταν ένα θέμα που αφορούσε μόνο την εφορία. Ε, εκείνη ήταν υπεύθυνη μόνο για τη φεργιότητα των ε, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και όχι για τη φορολογία. Ε, πήραν την απάντηση το 2015 όταν μια γερμανική τράπεζα, η Maple Bank, τότε ήταν θηγατρική μιας καναδικής τράπεζας, χρειάστηκε να κλείσει γιατί ακριβώς οι φορολογικές αρχές διεκδίκησαν ε, αχρεωστήτως καταβληθέντες ε, φόρους. Ε, τα, τα μέσα, τα χρηματοπιστωτικά που χρησιμοποιήθηκαν και οι άνθρωποι που διέπραξαν αυτά τα εγκλήματα ή που επέτρεψαν να διαπραχθούν αυτά τα εγκλήματα κάτω από την υποπτία των εποπτικών τραπεζικών αρχών όλα αυτά έγιναν λόγω του ότι οι νόμοι που παραβιάστηκαν ήταν νόμοι περί φορολογίας. Πώς μπορείς να ελέγξεις αν οι, οι διευθυντές των τραπεζών είναι σωστοί αν δεν προσπαθείς να ανακαλύψεις ε, οικονομικά εγκλήματα που διαπράττονται μέσα στις ίδιες τις τράπεζες. Τώρα, οι αρχές που μπορούν να εμποδίσουν εγκαίρω αυτού του είδου τα εγκλήματα είναι οι επόπτε των χρηματοπιστωτικών αγορών. Το νέο τρίκ ADR ανακαλύφθηκε πρώτα από την αρχή την Αμερικανική, την αντίστοιχη, την SEC και όχι τις γερμανικές φορολογικές αρχές. Η Buffin θα μπορούσε να έχει ανακαλύψει αυτή την υπόθεση με τα δεδομένα που είχε στη διάθεσή τη. Καταρχά ένας ε, πληροφοριοδότης έδωσε σχετικές πληροφορίες το 2007, αλλά έμεινε αναπάντητη η καταγγελία αυτή. Δεύτερον, η Μπαφίν θα μπορούσε να είχε δει τον μεγάλο εμπορικό όγκο που προκαλούσαν τα κουμ 6 μόνο ε, εξετάζοντας τον, τον όγκο καθημερινών συναλλαγών που ήταν πολλαπλάσιος από ό,τι τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου. Αναζητώντας το λόγο για μια τέτοια τεράστιο όγκο θα είχε ανακαλύψει και τα κουμ εξ και τα κουμ κουμ. Η αντίληψη του επόπτη Μπάφιν είναι αυτή στην οποία οφείλεται αυτή η τεράστια ζημιά για το γερμανό φορολογούμενο. Ότι δηλαδή δεν είναι υπεύθυνοι ε, όταν παραβιάζονται τέτοιου είδου νομοθεσίε. Μάθαμε στην ε, κοινοβουλευτική μα έρευνα ότι η Μπάφιν, ο γερμανό Επόπτη, δηλαδή δεν ενημερωνόταν από τις διάφορες ε, προσπά... για τι διάφορε προσπάθειε που έκανε το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει τα κουμέξ. Άρα λοιπόν συνέχισαν να εγκρίνουν τη δημιουργία επενδυτικών ταμείων που είχαν δημιουργηθεί μόνο και μόνο για την πώληση ε, την δόλια πώληση ε, των κουμέξ. Να χρησιμοποιήσω μια σύγκριση. Η Μπάφιν θα μπορούσε να έχει σταματήσει τους εγκληματίες εμποδίζοντας την αγορά του όπλου ε, με το οποίο δεν πράχθη ο φόνος. Σύμφωνα με την αρχές ε, που θεσπίζουν την ΕΣΠΑ, την, ε, τον Ευρωπαϊκό Φύλακα ε, για την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, δημιουργήθηκε τότε με στόχο να ελέγχει την ακαιρεότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών είναι πολύ πιθανό ε, και ε, μετοχές ασφαλιστικών εταιριών της Γερμανίας να χρησιμοποιήθηκαν σε δραστηριότητες κουμέξ και κουμ ε, <clears throat> Υπάρχει δηλαδή εδώ ρόλος και για τους επόπτες των ασφαλίσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με τη δική μας έρευνα, ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιριών δεν μπορούσε να καλυφθεί. Ελπίζω πως η ΙΟΠΑ θα μπορέσει να το ελέγξει αυτό. Να πω κάτι ακόμα. σημαντικέ πληροφορίε για την αποκάλυψη του σκανδάλου Κουμέξ, όπω και για τα υπόλοιπα μεγάλα φορολογικά σκάνδαλα, όπω τα Panama Papers και τα Lux Leaks, οι πληροφορίε δόθηκαν στι αρχέ και στου εισαγγελεί από του διάφορου πληροφοριοδότε. Αυτό δείχνει πόσο σημαντική είναι αυτή οι γενναίοι άνθρωποι στην καταπολέμηση του εγκλήματο. Για να στηριχθούν και να ενθαρρυνθούν οι άνθρωποι για να προβαίνουν σε τέτοιε καταγγελίε και να δίνουν τέτοιε πληροφορίε, χρειάζονται ε, συστήματα προστασία συνάδελφοί σας στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων αγωνίζονται γι' αυτό. Δυστυχώς στην Γερμανία ε, γίνονται ε, προσπάθειες να εξαιρεθούν οι λογιστές, οι φορολογικοί σύμβουλοι από τέτοιου είδους προστασία. Αυτά είχα σας να, πω και, να σας πω και ε, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ θα παραμείνετε μαζί μας σε απευθεία σύνδεση μέχρι τις 8 και τώρα ο κύριος Σπέγγελ. Ο καθηγητής κύριος Σπέγγελ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την πολύ ευγενική πρόσκληση που μου απευθύνατε και καθώς ε, το ζήτημα είναι πολύ τεχνικό και εξειδικευμένο από νομική άποψης, θα μιλήσω γερμανικά. Μιλάμε για το dividend stripping, δηλαδή χρηματιστηριακές συναλλαγές, γύρω από την ημερομηνία καταβολής διανομής των μερισμάτων, κατά τις οποίες ε, μετοχε, ε, πολλούνται μετοχές με ε, ε αξίωση μερίσματα, δηλαδή κουμ, και οι οποίες παραδίδονται στους αγοραστές τους είτε με είτε χωρίς ε, αξίωση διανομής. x στην ε, δημόσια αντίληψη πολλές φορές ε, αυτές οι, αυτές οι δύο, αυτά τα δύο είδη συχαίονται. Γι' αυτό και εγώ θα μιλήσω από κοινού και για τα δύο είδη. Θα ε, περιοριστώ και θα επικεντρωθώ στην κατάσταση της Γερμανίας. Αν έχετε ερωτήσεις για την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος, είμαι στη διάθεσή σας. Οι συναλλαγες κουμ CUM-X μαζί με τις ανοιχτές πωλήσει επιτρέπονταν στη Γερμανία στο 2011 και οδήγησαν ε, ο φόρος ε, των κερδών από κινητές αξίες να επιστρέφεται ε, πολλές φορές. Αυτό γινόταν μέσω της πολλαπλής βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας για τα κεφάλαια αυτά, για τα κέρδη αυτά. Γι' αυτό και μιλώ στην ουσία για φορολογική ληστεία. Η, αυτή, η δυνατότητα αυτή για την πολλαπλή επιστροφή ε, φορολογικών ε, ε, αξιών γινόταν μέσω της πολλαπλής βεβαίωσης. Παρακρατούνταν δηλαδή ο φόρος αυτός από τις διανέμουσες εταιρείες, βεβαιωνόταν από τις αποθεματικές τράπεζες των κατόχων, των μετόχων. Και έτσι εκδίδονταν δύο βεβαιώσεις, η μία που αφορούσε τον κάτοχο των μετοχών, κάτι που ήταν νόμιμο, και δεύτερον ε, για μια δεύτερη βεβαίωση για τον ε, προβαίνοντα ανοιχτή αγορά. Αυτή η δεύτερη βεβαίωση ήταν παράνομη, κάτι που έχει επιβεβαιωθεί και μέσα από πολλές ε, δικαστικές αποφάσεις. Για τις φορολογικές ζημίες ευθύνονται ο, ο ανοιχτός πολιτής ή οι αποθεματικές τους τράπεζες. Στη Γερμανία, λοιπόν, δεν υπήρχε ποτέ νομικό κοινό στην πραγματικότητα. Υπήρχε ε, μια παραβίαση συστηματική ε, τεχνικής φύσεως. Με βάση τις εκτιμήσεις μας, είχαμε φορολογικές απώλειες για την περίοδο 2005-2011 τουλάχιστον 7,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό είναι ο πιο συντηρητικός ε, υπολογισμός. Γιατί τα δεδομένα δυστυχώς είναι λυπή που έχουμε στη διάθεσή μας. Το 2012 ε, αναιρέθηκε αυτή η παραβίαση του συστήματος και πλέον ο φόρος ε, των κερδών από κινητές αξίες παρακρατείται από τις αποθεματικές τράπεζες και μόνο εκείνες μπορεί, μπορούν να βεβαιώνουν ε, την φορολογική αυτή παρακράτηση. Πώς ε, οδηγηθήκαμε σε αυτό το σκάνδαλο. Με το θέμα αυτό ασχοληθήκαμε το 2016-2017 στο Γερμανικό Κοινοβούλιο μέσω Εξεταστικής ε, Επιτροπής και τα αποτελέσματα, τα πορίσματα της Επιτροπής είναι πραγματικά συνταρακτικά. Υπήρξε ένα μείγμα από ε, πολιτική ανευθυνότητα, ε, ελλείψεις στους ελεκτικούς μηχανισμούς, αλλά και διασυνδέσεις με λόμπι. Η... Αυτό βεβαιώνεται και από το γεγονός ότι χρειάστηκαν πάνω από 10 χρόνια για να αναιρεθούν αυτές οι παραβιάσεις. Ε, μόλις το 2002 ενημερώθηκε ε, επισήμως η γερμανική κυβέρνηση. Και τα στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι και σήμερα ε, δεν ε, έχει καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί μαθηματικά, αριθμητικά το, το ύψος της φοροδιαφυγής αυτής. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι από τα έγγραφα ADR δεν προσδιορίζονται καθόλου ε, οι φορολογικές απώλειες, ζημίες του γερμανικού κράτους. Επίσης, το Υπουργείο, Γερμανικό, το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας φαίνεται ότι είχε ιδιαίτερες σχέσεις με την, ε, τράπεζα ε, με την Ένωση Γερμανικών Τραπεζών. Και τέλος, το 2009 Υπήρξε και μια εσφαλμένη εκτίμηση του Υπουργείου Οικονομικών που διευκόλυνε μάλιστα τις συναλλαγές Κουμέξ στη Γερμανία. Δεν αρκούν όμως όλα αυτά. Μέχρι σήμερα και εδώ και σχεδόν 40 χρόνια στη Γερμανία οι συναλλαγές κουμ-κουμ επιτρέπονται. Και αυτές βασίζονται στο ότι ε, πολίτες ή ταμεία που δεν έχουν την έδωση στη Γερμανία, λίγο πριν την διανομή των κερδών, των μερισμάτων, πουλούν τις μετοχές τους και αμέσως μετά την καταβολή των μερισμάτων τις ξαναγοράζουν. Ποιο είναι το κίνητρο. Υπάρχει ένα, ένα κενό στο φορολογικό δίκαιο. Διότι οι φορολογούμενες, ε, τα φορολογούμενα κέρδη ε, μετατρέπονται σε κινητές αξίες και έτσι επιστρέφεται ο φόρος ε, ε, κερδών από κινητές αξίες. Δεν είναι περσέ παράνομες αυτές οι συναλλαγές, όμως αντίκυνται στο πνεύμα του φορολογικού δικαίου. Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά θα έπρεπε να είχαν τουλάχιστον ελεγχθεί από το 2001. Οι δικές μας εκτιμήσεις για τις φορολογικές απώλειες για την περίοδο 2001 έως 2016 ε, κινούνται σε επίπεδα 5 έως 80 δισεκατομμύρια ε, ευρώ. Το Υπουργείο Οικονομικών, μάλιστα, στο, ε, έπειτα από κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, απαντούσα με ψευδή στοιχεία και το 2016 ε, ήθελε μάλιστα ακόμη και να ξεπλύνει αυτές τις συναλλαγές. Σε ό,τι αφορά το παρελθόν, το νομικό πλαίσιο εξακολουθεί να είναι ασαφές. Επιτρέπονται ακόμη αυτές τις συναλλαγές γιατί ακριβώς δεν έχει κλείσει αυτό το, κοινό, το κενό. Τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε μια λειτουργική διακυβέρνηση των ε, οικονομικών αρχών για να αποκαλύπτονται τέτοιου είδου σκάνδαλα, χρειαζόμαστε επίση ανταλλαγή απόψεων, ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για τα στοιχεία ε, για τον φόρο κερδών κινητών αξιών. Χρειάζονται διευρυμένε αρμοδιότητε για τι διοκτικέ αρχέ στην Ευρώπη σε φορολογικά ζητήματα και πρέπει επίση να συζητήσουμε για την ε, εύρυθμη λειτουργία Τη ε, αγορά της Ευρώπης, διότι αυτές οι συναλλαγές πολλές φορές πραγματοποιούνταν ε, σε διάφορες χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελευταίος ο θα είναι ο κύριος Σχέμ, Όμω όλοι οι προσκεκλημένοι ε, θα είναι διαθέσιμοι για ερωτήσεις, καθώς και ο κύριος Σαλεύσκη, δημοσιογράφο. Κύριε Σχέμ, έχετε το λόγο. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί ευρωβουλευτέ. Είμαι αρχισυντάκτη ε, του Κορεκτίβ Δημοσιογραφικού Οργανισμού και έχουμε ασχοληθεί με τα κουμ. Έχουμε 40 δημοσιογράφους ε, από 19 μέσα ενημέρωση σε 12 χώρες και εργαστήκαμε πάνω από 9 μήνες για να αποκαλύψουμε τη μεγαλύτερη φορολογική απάτη στην ιστορία της Ευρώπης. Οι ζημιές ε, ανέρχονται σε τουλάχιστον 55,2 δισεκατομμύρια ευρώ πώς ε, φτάσαμε σε αυτές ε, τις ε, αποκαλύψεις. Το 2017 είχαμε ήδη αποκαλύψει ότι από το 2001 ως το 2016 μέσω των συναλλαγων κουμ CUM-X και CUM-CUM είχαν προκληθεί ζημιές τουλάχιστον 31,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όμως, ήδη, ο κύριος Κρίστοφ Σπέγγελ ήδη είχε εξετάσει το θέμα αυτό. Μετά όμως το θέμα το πρόβλημα αυτό εξαπλώθηκε και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ε, όπως είπα, διεξήχθη μια έρευνα 9 μηνών και μας εξέπληξαν τα αποτελέσματα. Με, εκτός από τη Γερμανία, τουλάχιστον 11 χώρες ε, αφορά το ε, σκάνδαλο Κουμέξ. Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, κάτω χώρες Βέλγιο, Αυστρία, Δανία, ε, Ελβετία, Φιλανδία, Νορβηγία και Σουηδία. Όπως ε, είπα προηγουμένως, η συνολική ζημία σύμφωνα με την έρευνά μας ανέρχεται σε τουλάχιστον 55 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό προκύπτει τόσο από στοιχεία που έχουμε λάβει από φορολογικές αρχές όσο και από τις αναλύσεις μας ε, ε, δεδομένων της αγοράς τα ακριβή ποσά ε, έχουν ε, ω εξή. Μόνο για λίγε χώρε γνωρίζουμε τι ακριβώ έχει γίνει. Για τη Γερμανία η ζημία ανέρχεται στα 31,8 δισεκατομμύρια, για τη Γαλλία στα 17 δι, για την Ιταλία στα 4,5 δι, Δανία 1,7 και Βέλγιο 201 εκατομμύρια ευρώ. Ε, για τις υπόλοιπες ε, χώρες που αφορά το σκάνδαλο Κουμέξ δεν υπάρχουν ε, αξιόπιστα στοιχεία. Στην Γερμανία από το 2012 απαγορεύονται οι συναλλαγές Κουμέξ και από το 2016 οι συναλλαγές Κουμ Κουμ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας όμως συνεχίζουν να λαμβάνουν χώρα τέτοιου τύπου συναλλαγές. Είναι μεταλλάξεις των Κουμέξ και μάλιστα πολύ πιο επιθετικές και οι συναλλαγές αυτές είναι σε γενικές ε, γραμμές πολύ χειρότερες. Τι γίνεται, ε, διότι αφορούν ε, για παράδειγμα συναλλαγές με τα ADR. Τι γίνεται όμως στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν παραλλαγές των κουμ 6 που χρησιμοποιούνται ακόμα οι τράπεζες και οι traders συνεχίζουν να κάνουν πλιάτσικο στα δημόσια ταμεία. Η απάντηση είναι θετική. Ναι, ακόμα γίνονται τέτοιου τύπου συναλλαγές. Αυτό αποκάλυψε η μυστική μας έρευνα που προετοιμάζαμε εδώ και μήνες και μάλιστα το Σύμφωνα με το πόρισμά μας, ε, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Νορβηγία, η Φιλανδία, η Πολωνία και η Τσεχία είναι χώρες στις οποίες ακόμα και τώρα ε, γίνονται τέτοιου τύπου συναλλαγές ε, που κατακλέβουν τα δημόσια ταμεία. Αυτή η κλοπή λοιπόν συνεχίζεται σε όλη την Ευρώπη. Τι μπορούμε να κάνουμε. Στη Γερμανία αυτή τη στιγμή διεξάγεται μια συζήτηση για το αν θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση καταγγελίας ε, τέτοιας επιθετικής ε, φορολογικής ε, συμπεριφοράς. Οι φοροτεχνικοί, οι ελεκτές, οι ορκωτοί λογιστές θα ήταν λοιπόν υποχρεωμένοι αν υπήρχε τέτοια νομοθεσία να δηλώνουν τέτοιες περιπτώσεις όπου εντοπίζονται κενά στο φορολογικό δίκαιο. Ε, επίσης, θεωρώ πως η ε, δημοσιογράφοι η τέταρτη εξουσία έχει κάνει το έργο της. Τώρα η σκητάλη βρίσκεται σε εσά, αγαπητοί ευρωβουλευτές. Εμείς ε, οι δημοσιογράφοι έχουμε ήδη επισημάνει ότι υπάρχουν διάφορες παραλήψεις και διάφορες περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας από τις ε, από τους, ε, τις κρατικές αρχές ή τους ε, θεσμούς. Στην Γερμανία η... από τη στιγμή που έγιναν παράνομες οι συναλλαγές κουμεξ και κουμ δεν σταμάτησαν βέβαια μετατοπίστηκαν και πήγαν πιο βόρεια, πήγαν στη Δανία. Για μένα πρόκειται για εγκληματική συμπεριφορά, εγκληματική παρέμβαση στα δημόσια οικονομικά. Η Ευρώπη χρειάζεται να βρει έναν κοινό δρόμο, να αντιμετωπίσει από κοινού την κατάσταση και αυτό προϋποθέτει τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αρχής. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η Ευρώπη χρειάζεται ένα οικονομικό FBI και μάλιστα αμέσως. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε τώρα στην ανταλλαγή απόψεων με τους ε, ευρωβουλευτές. Γνωρίζετε τους κανόνες. Ο καθένας σας έχει... Ε, μάλλον έχετε όλοι πέντε λεπτά χρόνο, το πολύ δύο λεπτά ο καθένας. Γι' αυτό λοιπόν Φροντίστε να είστε σύντομα και περιεκτικοί και μην ξεχνάτε ότι ο προσκεκλημένος μας από το Γερμανικό Κοινοβούλιο θα πρέπει να φύγει στις 8. Θα ξεκινήσουμε με τους ε, κεφαλής των ε, πολιτικών ομάδων και μετά θα περάσουμε σε όσους έχουν ζητήσει το λόγο. Πρώτος ομιλητής είμαι εγώ. Θα ξεκινήσω λοιπόν με τις δικές μου ερωτήσεις Έχω δύο ερωτήσεις. Η μία αφορά τα cum και η άλλη τα CUM-CUM. Σχετικά με τα cum αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πώς γίνεται τον 21ο αιώνα να ζούμε τέτοια κατάσταση. Ε, τα μερίσματα διανέμονται μόνο μία φορά. Πώ πώς είναι λοιπόν ε, δυνατόν να μην μπορούμε να διαπιστώσουμε σε πόσους έχουν διανεμηθεί οι μερίσματα και πόσοι έχουν λάβει αυτά τα πιστοποιητικά. Οι φορολογικές αρχές ε, μάλιστα δεν μπορούν να διαπιστώσουν ε, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης ενός τίτλου. Εξηγήστε μου λοιπόν πώς ε, είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο σε ό,τι αφορά την επιστροφή φόρου. Επίσης, Είναι αυτή η πρακτική η ίδια με αυτό που λέμε dividend washing, ξέπλυμα μερισμάτων. Είναι δηλαδή μια συναλλαγή που έχει ακριβώς, αυτό, ακριβώς αυτόν τον σκοπό. Παρακαλώ επιβεβαιώστε. Και επίσης η πρακτική αυτή ε, χρησιμοποιείται από αυτές ε, μόνο τις ε, χώρες ή θεωρείται νόμιμη γενικότερα. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου και σας παρακαλώ να μην ξεπεράσετε τα πέντε λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, θα απαντήσω και θα απαντήσω στα αγγλικά, γιατί είναι πολύ τεχνικό το θέμα. Πρώτη ερώτηση. Πώς είναι δυνατόν να εκδοθούν δύο φορολογικά πιστοποιητικά για, έγγραφ, για μετοχές αυτό έχει να κάνει με το χρόνο και μόνο. Την ημέρα την κατά την οποία εμπορεύονται αυτές οι μετοχές και την ημέρα την οποία γίνεται η αγοροπολισία. Ε, για παράδειγμα, στην Γερμανία αυτό το χρονικό περιθώριο είναι δύο μέρες. Για κάποιες άλλες χώρες όμως ε, είναι τρεις ημέρες κατά τις οποίες καταβάλλονται τα μερίσματα. Τότε λοιπόν λαμβάνουν χώρα αυτές οι συναλλαγές ο νόμιμος ιδιοκτήτης των μετοχών την ημέρα της καταβολής ε, μερισμάτων λαμβάνει το μέρισμα και το πιστοποιητικό που εκδίδει η ε, τράπεζα θεματοφύλακας. Αυτό μέχρι εδώ καλά. Τώρα, οι συναλλαγές ε, σε μετοχές έχουν γίνει με μέρισμα, cum dividend, όμως η συνέχεια γίνεται χωρίς, η πώληση γίνεται χωρίς μέρισμα την ημέρα που καταβάλλεται. Αυτό ε, οδηγεί στο εξή. Εκείνος που προβαίνει σε ανοιχτή αγορά πληρώνει στην ουσία ε, ένα πλασματικό, ένα κατασκευασμένο μέρισμα, το οποίο δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου μερίσματος παρά το γεγονός ότι η αποθεματική τράπεζα έχει εκδώσει και άλλα πιστοποιητικά ε, σύμφωνα με τα οποία δεν γνωρίζουν αν η πληρωμή αφορά ένα πραγματικό μέρισμα ή ένα πλασματικό. Αυτό το παραθυράκι ήταν τεχνικής φύσης και υπήρχε στην Γερμανία και τη Δανία. Το 2012 σταμα... έκλεισε στη Γερμανία, διότι τώρα, τώρα η ίδια τράπεζα είναι εκείνη που... Ε, συλλέγει τα, ε, και διανέμει τα μερίσματα και ε, εκδίδει τα πιστοποιητικά. Τώρα, γιατί χρειάστηκε πάνω από 10 χρόνια για να κλείσει αυτό το τεχνικό παραθυράκι. Καλή ερώτηση. Τώρα, ε, σε ό,τι αφορά την ερώτηση για τα κουμ-κουμ, είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα. Γίνεται αυτό το stripping, dividend stripping, και το παραθυράκι στη Γερμανία δεν έχει κλείσει ακόμα γιατί οι πληρωμές ε, μερισμάτων, σε μη ε, φορολογικούς ε, κατοίκους δεν είναι δυνατή. ενώ η, όταν αλλάζουν χέρια υπάρχει τέλος παρακράτησης φόρου. Ευχαριστούμε για τις εξηγήσεις. Δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικά αυτά. Για τους σοσιαλιστές η Ο Πέτερ Σίμωρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Είμαστε και οι δύο από το Μανχάιμ, οπότε ε, νομίζω ότι θα συνεννοηθούμε και στα γερμανικά. Το ερώτημα μου απευθύνεται σε εσά. Είπατε πόσο δύσκολο είναι να προσδιορίσει κανείς ε, χρηματικά τα ποσά. Είπατε ε, ο συνάδελφός σας ότι έχει καταλήξει στα περίπου στα 55 δισεκατομμύρια. Εσείς μπορείτε να μας πείτε πώς, ποια μεθοδολογία ακολουθήσατε, ποια μεθοδολογία υπολογισμού ε, ακολουθήσατε για να φτάσετε στους δικούς σας ε, αριθμούς. Όταν ούτε η ίδια η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας δεν φαίνεται να μπορεί να συλλέξει αυτά τα τόσο πολύ σημαντικά στοιχεία. Δεύτερο ερώτημα για τον κύριο Σπέγγελ. οι μεγάλες συμβουλευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται πάντοτε σε αυτά τα πολύ μεγάλα φοροτεχνικά ζητήματα, οι Big Four εταιρείες, ε, έχουν κάποια διασύνδεση είτε με την ανάπτυξη είτε με την ε, αγοραπολισία τέτοιων ε, προϊόντων τέτοιων, με αυτές τις χρηματιστηριακές συναλλαγές. Και κάτι τελευταίο. Έχω μιλήσει με πολλά μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και μου έχουν πει ότι η ευρωπαϊκή διάσταση δεν συζητήθηκε καθόλου στο Bundestag γιατί θεωρήθηκε ότι ήταν αδύνατον να υπάρχει και ευρωπαϊκή διάσταση. Ότι στη χειρότερη περίπτωση θα μπορούσαν ενδεχομένως να είχαν υπάρξει ε, κάποιες, κάποιες δευτερεύουσα σημασίες επιπτώσεις σε άλλες χώρες. Μπορείς να μας πεις ε, λίγο περισσότερα στοιχεία ως προς αυτό. Ευχαριστώ. Τρία λεπτάκια έχουμε για την απάντηση παρακαλώ. Στα γερμανικά. Ζήμων, κύριε Ζήμων. Για τις ζημίες που προήλθαν από το σκάνδαλο QM, QMX. Εμείς λάβαμε δεδομένα από, από την εταιρεία Clearstream που διαχειρίζεται τις χρηματιστηριακές συναλλαγές στο γερμανικό χρηματιστήριο. Μας έδωσε στοιχεία για το 2005-2011 και στη βάση αυτή προσδιορίσαμε ανοιχτέ πωλήσει και με βάση αυτό το στοιχείο καταλήξαμε στο, ε, στη φορολογική ζημία 7,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για αυτή την περίοδο. Γνωρίζοντας όμως ότι τέτοιες συναλλαγές cum-ex γίνονταν στη Γερμανία ήδη από τα τέλη της, ε, της δεκαετίας του 90 και γι' αυτό αυτόν ακριβώ το λόγο πρόκειται για τον πλέον συντηρητικό υπολογισμό. Για, τα, για τις συναλλαγές κουμ-κουμ ε, συνυπολογίσαμε τις διανομές μερισμάτων ε, του DAX, των εταιριών που συμμετέχουν στο DAX για την περίοδο 2001-2016. Τα στοιχεία αυτά υπάρχουν. Και θεωρήσαμε ότι όλε οι συμμετοχέ που δεν ανήκαν σε γερμανικά συμφέροντα, σε γερμανικά χέρια, ε, προέβαιναν σε τέτοιε συναλλαγέ. Αν δεν υπάρχει ε, συμφωνία ε, αποφυγής διπλής Ε, μιλάμε για 25% του, του φόρου. Στα 15% φόρος εισοδήματος το μέγιστο, η μέγιστη ζημία ανέρχεται στα 50 περίπου δισεκατομμύρια. Αν μιλάμε για 25% ε, φόρο ε, εισοδήματος επί κερδών, ε, μιλάμε για 80%, για 80 εκατομμύρια. Γι' αυτό, με αυτόν τον τρόπο δηλαδή, καταλήξαμε, για τα κουμέξ είναι περίπου 7 δισεκατομμύρια. Μου είπαν οι συνάδελφοι ότι το 50 με 80 στο οποίο καταλήξαμε για το κουμκουμ είναι λίγο πολύ για να ισχύει, οπότε παίρνουμε περίπου το μισό, δηλαδή γύρω στα 32 δισεκατομμύρια θεωρούμε ότι είναι μια πολύ πιθανή ζημία αυτή που προκλήθηκε. Να συμπληρώσω κάτι κι εγώ. Λόγω αυτή τη υπόθεση εργασία, αυτό που είπατε δηλαδή ότι όλε οι συναλλαγέ με το εξωτερικό έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευση, ε, ε, γι' αυτό συντηρητικά είπαμε ότι μάλλον όχι 100% αλλά ας πούμε οι μισές συναλλαγές να χαρακτηρίζονταν ή να εντάσσονταν σε αυτά τα συστήματα CUM-X και κάπως έτσι καταλήξαμε σε αυτό το 32 δισεκατομμύρια ε, ευρώ. Κύριε Σικ, θέλετε να απαντήσετε γιατί νομίζω ότι απευθυνθήκε ένα ερώτημα και σε εσά. Ναι, για, τους, ε, για τις συμβουλευτικές εταιρείε και τις φοροτεχνικές εταιρείε και τον ρόλο τους. Είναι αλήθεια ότι τα διοικητικά συμβούλια επενδυτικών και τραπεζικών ιδρυμάτων είχαν πάντοτε πολύ καλή νομική προστασία και εξασφάλιση ε, με εξαιρετικά ε, εξειδικευμένες ε, νομικές συμβουλές που λάμβαναν από αντίστοιχα εξειδικευμένες νομικές φοροτεχνικές εταιρείες. Γι' αυτό και εμφανίζονταν ως νόμιμες οι συναλλαγές και οι δραστηριότητες αυτές. Ε, δεν ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με τις τέσσερις μεγάλες λογιστικές εταιρείες. Ούτε καταφέραμε να προσδιορίσουμε, ούτε βεβαίως και να συζητήσουμε, να αναλύσουμε τον ρόλο αυτών των τεσσάρων εταιρεών. Ε, Η αλήθεια είναι πάντως ότι όπως και στην οικονομική κρίση ε, ούτε σε αυτό το θέμα ε, ε, στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Είπατε και για την Εξεταστική Επιτροπή του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Είναι αλήθεια ότι μάλλον υπήρξε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση με τον ομιλητή. Πρόεδρος, δεν υπάρχει εκπρόσωπος του ECR, είναι όμως εδώ ο κύριος Κλίνς από τους Φιλελεύθερους. Κάθε 7 χρόνια ασχολούμαστε εδώ με το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό ε, πλαίσιο και βλέπουμε ότι με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και γίνεται μάχη για κάθε ευρώ και όλα αυτά ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν σκάνδαλα διψήφιων, διψήφιων αριθμών δισεκατομμυρίων και φορολογική απάτη. Φανταστείτε δηλαδή τι γίνεται. Είναι πραγματικά καταστροφή. Γιατί, πώς οδηγηθήκαμε εδώ. Γιατί όπως ε, είχαμε πει και στη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 ε, υπάρχουν εγκληματικέ ενέργειες που ε, οφείλονται και στον, στην, στις αχόρταγες διαθέσεις διαφόρων κύκλων και εταιριών. Πώς θα τα ελέγξουμε όλα αυτά. Το ερώτημά μου το πρώτο είναι ποιο τελικά αποκόμισε κέρδη από αυτέ τι απάτε. Ήταν φοροτεχνικοί, οι τράπεζες, ήταν δικηγόροι, ήταν οι ίδιοι οι μέτογοι. Ποιο ήταν ο βασικό ωφελούμενο ή ήταν ένα μείγμα όλων αυτών. Ποιο ωφελήθηκε. Δεύτερον, δεν θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ανεξάρτητα από τις καταδικαστικές αποφάσεις που κάποια στιγμή φαντάζομαι ότι θα ληφθούν, ελπίζω τουλάχιστον, δεν είμαστε ε, υποχρεωμένοι να πούμε ότι όποιος έχει εμπλακεί σε τέτοιες ε, δραστηριότητες χάνει την άδεια άσκηση επαγγέλματό του. Ένας τραπεζίτης δηλαδή, που έχει συμμετάσχει με τον έναν με τον άλλο τρόπο σε τέτοιες δραστηριότητες, δεν πρέπει να πούμε ότι δεν επιτρέπεται να ξαναμπεί ε, σε αυτό το εμπόριο ε, και σε αυτές τις εναλλαγές. Αποτρε... Ως αποτρεπτικό μέτρο. Δεύτερον, ε, γίνεται λόγο πάντοτε για αυτά τα short sale, τι ανοιχτέ πωλήσει και πολλοί λένε ότι αυτά είναι ε, πολύ σημαντικά για τη ρευστότητα, για τι αγορέ κτλ. Το ερώτημα μου είναι, είναι πραγματικά τόσο αναγκαίε αυτέ οι συναλλαγέ. Γιατί να μην τις περιορίσουμε αυτές τις ε, ανοιχτέ πωλήσει. Τι θα ήταν το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί. Τρίτον, πρόεδρος, συγγνώμη, αν κάνετε τόσο μεγάλες ερωτήσεις, απάντηση δεν πρόκειται να πάρετε. Ωραία. Εντάξει, τότε δεν θα πω κάτι για τη διακυβέρνηση που ήθελα. Θα πω όμως κάτι τελευταίο. Στους φόρους γνωρίζουμε ότι η φορολογική πολιτική είναι εθνική αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει όμως να υπάρξει μια τουλάχιστον μερική εναρμόνιση των φορολογικών δεδομένων και φορολογικών πολιτικών ώστε να σημειώσουμε την οποιαδήποτε πρόοδο που θα μπορούσαμε να σημειώσουμε. Θα μοιραστούμε το χρόνο για τις απαντήσεις. Καταρχάς, ε, ποιο αποφελήθηκε, όλοι όσοι αναφέρατε, τράπεζες, ε, δικηγόροι, φοροτεχνικοί, επενδυτές, μην ξεχνάμε, εύποροι ε, πολίτε οι οποίοι είναι σε θέση να επενδύσουν τεράστια ποσά σε αυτές τις συναλλαγές και να αποκομίσουν και τεράστια κέρδη. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας που μένει εκτό. Τώρα, απαγόρευση άσκηση επαγγελματο. Νομίζω ότι πρέπει να έρθει καιρός και γι' αυτό. Όταν θα γίνουν οι πρώτες ε, δίκες και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, τότε θα είναι και κάτι αναμενόμενο να γίνει απαγόρευση άσκηση επαγγέλματο. Όμω αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσουν οι επαγγελματικέ ενώσει. Ναι, ε, θα συμφωνήσω κι εγώ σε αυτό. Τώρα, ανοιχτές πωλήσει, πώς μπορούμε να διαχειριστούμε όλες αυτές ε, τις ε, συναλλαγές, δανεικές μετοχές κτλ. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε καταχρήσεις και φορολογική απάτη. Νομίζω πως εδώ το θέμα είναι στα κίνητρα, τα φορολογικά κίνητρα, να καλύψουμε τα κενά μέσω να κλείσουν τα παραθυράκια μέσω της ε, νομοθεσίας, μέσω αποτρεπτικής ε, νομοθεσίας. Στις ανοιχτές ε, πωλήσει ακούσαμε τι συμβαίνει, ειδικά την εποχή της ψηφιοποίησης είναι δυνατόν να κλείσουμε όλα τα παραθυράκια για να μην υπάρχει κάτι που θα μας ξεφύγει. Τώρα, όλο το σύστημα της ε, συλλογής ε, φόρου κινητών αξιών θα πρέπει να επανεξεταστεί. Αυτό βέβαια δεν είναι το θέμα μας τώρα. Στην Ευρώπη όμως εκτιμούμε ότι κάθε χρόνο χάνονται 150 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω τέτοιων ε, συναλλαγών και πρακτικών. Το θέμα είναι να κλείσουμε αυτά τα κενά τα οποία είναι ανοιχτά εδώ και χρόνια, τα οποία εκμεταλλεύονται ε, όλοι όσοι επωφελούνται από αυτό. Και αυτό είναι προς όφελος όλων των κρατών μελών. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής εκ μέρους της ΕΚΟΥ, ο κύριος Παδημούλης Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζήτησα στην προηγούμενη Ολομέλεια τον Νοέμβριο να συζητήσουμε το θέμα και στην Ολομέλεια και χαίρομαι που ξεκινάει και η εξέταση του εδώ με τη συμβολή ειδικών. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σπέγγελ μας είπατε ότι το θέμα θα μπορούσε αυτό το γιγαντιαίο σκάνδαλο, αυτή τη φορολογική απάτη, να έχει ελεγχθεί από το 2001, αντί για αυτό το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας έδινε ψευδή στοιχεία και πήγε και το 2016 να το κουκουλώσει. Θα ήθελα να μας πείτε λεπτομέρειες. Ποιοι, πότε και πώς. Ε, και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σρόμ που μας είπε ότι το πλιάτσικο συνεχίζεται ακόμη σε αρκετές χώρες. Αν μπορεί να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Και η τρίτη μου ερώτηση για το πώς μπορούν να κλείσουν αυτές οι τρύπε που επιτρέπουν αυτό το γιγαντιαίο έγκλημα της φορολογικής απάτης αρκετών πλουσίων ανθρώπων σε βάρος των δημόσιων ταμείων και των συνεπών φορολογουμένων, που είναι πολύ πιο φτωχοί από αυτούς αυτό που λέτε ένα οικονομικό ευρωπαϊκό FBI. Θα μπορούσατε κύριε Στρόμ να μας το περιγράψετε. Χρειάζεται ευρωπαϊκές λύσεις και ισχυρότερους ευρωπαϊκούς θεσμούς ελέγχου ή μπορούν και μόνα τους τα κράτη-μέλη να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε τις απαντήσεις παρακαλώ. Για το ερώτημά σας που απευθύνονται σε μένα. Από δημοσιογραφικούς κύκλους, πριν από 20 χρόνια περίπου, το 1997, εμφανίστηκαν οι πρώτες ενδείξεις για το ότι πραγματοποιούνται συναλλαγές κουμέξ στη Γερμανία. Το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας ενημερώθηκε από την ε, Ένωση Τραπεζών της Γερμανίας επίσημα, μέσω επιστολής, για το ότι πραγματοποιούνται τέτοιες συναλλαγές κουμέξ στη Γερμανία και ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σε σχέση με τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας για, τα κέρδη, για τους φόρους από ε, κέρδη από κινητές αξίες αλλά ταυτόχρονα συνοδεύτηκε από, από την επισήμανση ότι αυτό δεν μπορεί να λυθεί μόνο στο πλαίσιο μια ε, εθνική ένωμη τάξη, διότι ακριβώ επειδή οι συναλλαγέ αυτέ γίνονται σε πολλέ χώρε, αυτό το manufactured dividend, το μέρισμα που διανέμεται εκτός Γερμανίας, δεν είναι φορολογητέα ε, αυτά τα, τα μερίσματα στην Γερμανία. Αυτή την πληροφορία το Υπουργείο μας την έλαβε ε, το Δεκέμβριο του 2002. Το 2006-2007 έγινε τροποποίηση της νομοθεσίας και που κατέστησε την, τα μερίσματα ε, φορολογητέα, αλλά μόνο όταν αυτά διανέμονται από γερμανική τράπεζα. Όλες οι περιπτώσεις που έγιναν γνωστές στη Γερμανία όμως αποδεικνύουν ότι αυτές οι δραστηριότητες, συναλλαγές πραγματοποιούνται πάντοτε μέσω χωρών του εξωτερικού. Το 2012 έκλεισε το παραθυράκι αφού αναγνωρίστηκε ότι την απάτη μπορείς να την ε, καταπολεμήσεις μόνο όταν υπάρχει ένα, πιστοποιητικό από εκείνη την υπηρεσία που ε, τελικά αποδίδει το φόρο ε, στις φορολογικές αρχές της Γερμανίας. Αυτό είναι το ανησυχητικό, ότι χρειάστηκαν 10 χρόνια για να κλείσει αυτό το απλό παραθυράκι. Έγινε μια μυστική έρευνα, ολόκληρη επιχείρηση. Είχαμε επαφές στο Λονδίνο με διάφορους ε, traders και ε, είχαμε συζητήσει λοιπόν μαζί τους, είχαμε λάβει κάποια έγγραφα και παρατηρήσαμε ότι αυτού του είδους οι συναλλαγές διεξάγονται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις μας είχαν πει ότι να, αν, είχε, αν είχα επενδύσει αυτό το ποσό θα είχα ε, πολλαπλάσια κέρδη. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, το, την ανάγκη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού οργανισμού. Ε, νομίζω πως ε, όλα συνοψίζονται στο ότι χρειάζεται επικοινωνία, χρειάζεται ανταλλαγή πληροφοριών. Δεν γνωρίζω την φορολογική ε, νομοθεσία της Δανίας, δεν ξέρω ούτε καν τη γλώσσα, όμως έχω κάνει έρευνες εκεί, έχουμε κάνει ανταλλαγή πληροφοριών με τους συναδέλφους και Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να πάρει, για παράδειγμα, τηλέφωνο στην Ιταλία και να πεις «φέρτε μου τα στοιχεία». Να τα δω. Χρειάζεται ε, επικοινωνία, ενημέρωση. Δεν ε, θέλουμε επίσης ε, να είμαστε οι σερίφιδες που θα κυνηγούμε τους κακούς και θα μας σταματάνε στα σύνορα. Ε, και τότε θα εξαφανίζεται ο κλέφτη. Χρειάζεται ανταλλαγή ε, πληροφοριών, ε, έστω σε ένα ελάχιστο επίπεδο, σε ένα πολύ περιορισμένο επίπεδο και νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει βάση για να δουλέψουμε περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Σβέν Γκίγκολτ εκ μέρου των Πρασίνων. Σα ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να υποβάλω τις εξής ερωτήσεις, καταρχάς στον κύριο Σαλεύσκη, αλλά επίσης στον κύριο Σπέγγελ και στον κύριο να θέλουν να απαντήσουν. Μπορείτε να μας πείτε λεπτομέρειες όσο γίνεται πιο, με μεγαλύτερη ακρίβεια για το ποιο είδος ε, φορέων και αν θέλετε να τους κατονομάσετε, ε, κατονομάστε τους, αλλά ποιο είδους ε, φορείς συμπεριλαμβάνονταν σε αυτό την την υπόθεση σε διάφορες, ε, στα διάφορα κράτη. Ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες, ταμεία, τι είδου ταμεία, τι είδου σύμβουλοι, παρακαλώ να μας τα πείτε όσο γίνεται πιο ξεκάθαρα. Τι είδου φορεί λοιπόν ήταν αναμεμειγμένοι. Δεύτερον, αν δεν μπορείτε να τελειώσετε αυτό τον κατάλογο, μπορείτε να μα στείλετε ένα τέτοιο κατάλογο επί τη βάση των πληροφοριών που έχετε στη διάθεσή σα. Έπειτα, θα ήθελα να γνωρίζω και από τους τρεις σας ποιες, ποιοι νόμοι είναι αυτοί οι οποίοι παραβιάστηκαν σύμφωνα με τις ε, δικές σας πληροφορίες και πού και σε ποια ακριβώς σημεία, σε ποια κρατη έχουμε παραβίαση της νομοθεσίας. Τέλος, τον κύριο Σουμ, είστε έτοιμος να μοιραστείτε κάποιο από το υλικό που έχετε στη διάθεσή σας με το Ευρωκοινοβούλιο και υπό ποιους όρους. Ευχαριστώ. Και τώρα οι απαντήσει. Ευχαριστώ για τους φορείς ε, που συμμετείχαν σε αυτές τις δραστηριότητε. Θα μπορούσα να πω συνοπτικά το εξή. Όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα με τις διάφορες ιδιότητες που μπορεί να εμφανίζεται. Γιατί προφανώς κανείς χρειάζεται πολλά χρήματα για να κάνει τέτοιε συναλλαγέ. Μιλάμε για ιδιώτε επενδυτέ που έχουν τέτοια στη διάθεσή του ή ε, τράπεζε που έχουν βεβαίω τέτοια ίδια κεφάλαια ή τράπεζε που αντιστοίχω ε, δημιουργούν τέτοια φόν, τέτοια ταμεία ε, τα οποία μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιου είδου συναλλαγέ. Αυτή είναι ε, η βασική αρχή. Χρειάζεσαι ανθρώπου που έχουν πολλά χρήματα. Έπειτα όμω υπάρχουν και τράπεζε οι οποίε λένε ότι χορηγούσαν δάνεια χωρί να ξέρουν ακριβώ για, ποιον και για, για ποιο λόγο και σε ποιου τα έδιναν τα δάνεια αυτά. Φανταστείτε εσεί να πάτε να αγοράσετε ένα σπίτι. Δεν θα σα ρωτήσει η τράπεζα ποιο σπίτι ακριβώ θέλετε να αγοράσετε και τι χαρακτηριστικά έχει. Ε, Γι' αυτό ε, ε, έχουν σίγουρα ευθύνε πολύ μεγάλε οι τράπεζε. Από εκεί και πέρα ε, έχουμε και του μετόχου οι οποίοι δανείζουν, πολλούν, αγοράζουν τέτοιες ε, μετοχές συνεχώς και οι οποίοι πολύ εύκολα μπορούν να πούν, ε, να, πούν να ισχυριστούν ότι δεν, ήξερα, δεν, δεν, δεν γνώριζα όλες τις πληροφορίες. Ε, είναι λίγο περίεργο βέβαια που αυτές οι αγροπολισίες γίνονταν συνήθως γύρω από την ημερομηνία ε, της διανομή των μερισμάτων. Υπήρχαν επίσης και ε, νομικές εταιρείε, ασφαλιστικές εταιρείε, οι οποίες συνεργάζονταν για να ασφαλίσουν αυτές τις συναλλαγές. Και αυτό ε, ξέπλαινε, αν θέλετε, και νομιμοποιούσε τύπης τη διαδικασία. Υπάρχει λοιπόν μια πλειάδα παραγόντων φορέων που ωφελούνταν. Βεβαίω, βασική ε, κινητήρη μοχλή είναι ε, οι μέτοχοι. Εκείνοι που πραγματικά κατέχουν, αν θέλετε, αυτές τις μετοχές και που λαμβάνουν αυτά τα μερίσματα ή απαλλάσσονται από την σχετική φορολόγηση των, ε, των μερισμάτων. Και επειδή το ερώτημα επίσης ήταν αν μπορούμε και να κωδικοποιήσουμε όλα αυτά που σας λέμε. Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου και θα σας δώσω και κωδικοποιημένα τα σχετικά στοιχεία, αφού μου τα ζητήσατε. Μία υπόθεση θέλω να περιγράψω εγώ, την Δανέζικη, που ε, συζητείται αυτή τη στιγμή και εξετάζεται στο δικαστήριο στο, στο, δικαστήριο στο Λονδίνο ότι ε, δημιουργήθηκε ε, ένα σταξιδοτικό ταμείο ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε short sales ανοιχτή πώληση στη Δανία. Σε αυτή, τη, στην, σε αυτή δραστηριότητα συμμετείχε και μια πολύ, γερμανική, πολύ μικρή γερμανική τράπεζα το Mind και έλαβαν ένα φορολογικό βάουτσερ κουπόνι από τις δανέζικες αρχές στο ΜΑΙΝΤ και πήγαν ε, μετά με αυτό το βάουτσερ για να πάρουν ε, την επιστροφή φόρου από την Barclays στην Αγγλία και από αυτή την τράπεζα, από την Barclays, τα, τα χρήματα μεταφέρθηκαν στην τράπεζα Βάρεγκολ στο Αμβούργο και χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα αυτά για ξέπλυμα, για νομοποίηση παράνομων εσόδων. Βλέπετε δηλαδή ότι η κεφαλαία αγορά στην Ευρώπη οι ε, προβαίνοντες πολλές φορές σε τέτοιες ε, δραστηριότητες βρίσκονται εκτός Ευρώπης. Ε, εδώ είχε δημιουργηθεί ένα συνταξιδοτικό ταμείο στι ε, ΗΠΑ. Είναι πάρα πολύ αδιαφανέ το, το όλο σύστημα και συμμετέχουν πάρα, πάρα πολλοί ε, παράγοντε από διάφορε χώρε. Τώρα, αν ε, υπάρχουν και άλλε περιπτώσεις παραβίασης δικαίου. Τώρα, ξέρω την περίπτωση της Γερμανίας. Στη Γερμανία είναι, πρόκειται για απάτη, για φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή. Εκεί εστιάζουν οι αγωγές που έχουν γίνει. Πρόκειται για τραπεζίτες, για traders που έχουν συνεργαστεί, έχουν συνεννοηθεί έτσι ώστε να γίνουν αυτές οι συναλλαγές. Αυτό για μένα είναι οικονομικό έγκλημα και οργανωμένο έγκλημα μάλιστα. Να προσθέσω κάτι. Αυτή η συνεννόηση που χρειάζεται έτσι ώστε να γίνουν αυτές οι κυκλικές συναλλαγές είναι από μόνη της παράνομη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτοί οι traders ε, για να παρακάμψουν ε, τον ε, έλεγχο χρησιμοποίησαν Snapchat και μάλιστα όχι στα επαγγελματικά κινητά τους αλλά στα προσωπικά τους κινητά. Snapchat το οποίο ξέρετε πώς λειτουργεί μετά από λίγο ξεφανίζεται το μήνυμα για να μην αφήνουν ίχνη. Αυτό σύμφωνα με το βρετανικό δίκαιο είναι εγκληματική πράξη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μποργέζιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από τα στοιχεία από τις τρέχουσες έρευνες και από την εισαγγελία της κολονίας προκύπτει ότι σοβαρό έγκλημα έχει διαπραχθεί από τα τμήματα Investment Bank και Trading των εξή τραπεζών όσον αφορά τη Γερμανία. Σαταντέρ, Deutsche Bank, HCSB, ε, Goldman Sachs και Maygrid Bank. Δηλαδή, μας δίνει αυτή η έρευνα στοιχεία ότι ένα τέτοιο μεγάλο ε, σκάνδαλο, έγκλημα όπως μας είπαν ε, πραγματικά καλύπτει ένα τεράστιο κομμάτι της γερμανικής χρηματοπιστωτικής βιομηχανίας και αυτό κατέστη δυνατό μόνο και μόνο λόγω τεραστίων δυνατοτήτων πίστοσης από αυτές τις τράπεζες. Το πρώτο λοιπόν που θα πρέπει να μας προβληματίσει είναι το εξή και θέλω να το μοιραστώ με τους εμπειρογνώμενες μας. Αν αυτές οι μεγάλες τράπεζες ήταν υποχρεωμένες από κάποιο νόμο είδους ε, ε διαχωρισμού ανάμεσα στις εμπορικές τράπεζες και τις ε, απλές τράπεζες θα είχαν μπορέσει να προσφέρουν τις δυνατότητες αυτές και αυτές τις υπηρεσίες σε αυτά τα ταμεία και ε, να ε, έχουν αυτά τέτοια κέρδη. Πρέπει αυτό να το σκεφτούμε γιατί οι γερμανικές φορολογικές αρχές γνώριζαν τι συνέβαινε από το 2002 αλλά τότε διερωτώμεθα από αυτή τη τεράστια υπόθεση και όλες αυτές τις συναλλαγές που από ό,τι φαίνεται συμμετείχαν και μετοχές και από την Γαλλία και από την Ισπανία και από το Βέλγιο και από τη Δανία η Ευρωπαϊκή Εποπτεία τι κάνει τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που ασχολείται με τόση μεγάλη προσοχή να καθορίσει πράγματα και να ελέγξει πράγματα που είναι πολύ λιγότερο σημαντικά και όχι μόνο δεν κατάλαβε τι γινόταν, αλλά καθυστερεί και τόσο πολύ να δράσει. Δηλαδή, έχουμε την εντύπωση ότι γίνεται μια επιχείρηση συγκάλυψης αυτών των εγκλημάτων, που είναι πάρα πολύ σοβαρά αδικήματα. Και είναι εντυπωσιακό το επίπεδο της ε, έλλειψης προσοχής που έχει δοθεί από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν παρέμβει για μια τέτοια κατάσταση. Και όπως είπα, αποκαλύφθηκαν από ε, παράγοντες εξωτερικούς της Ένωσης. Η απάτη όλη αυτή συνεχίζεται δε, όπως μας λένε οι εμπειρογνώμονες, με νέες μορφές, χωρίς να έχει γίνει επιτυχώς ε, προσπάθεια να διακοπεί όλη αυτή η κατάσταση. Ποιος θα ήθελε να απαντήσει. Ποια ήταν η ερώτηση ακριβώς, παρακαλώ. Ε, άκουσα μια δήλωση, αλλά καμία ερώτηση. La demanda era implicita. Μα η ερώτηση ήταν ε, την υπονόησα, δηλαδή από τη δική σας εμπειρία και μέσα από την έρευνά σας, ε, τι συγκεκριμένα δεν λειτουργήσε σε επίπεδο ευρωπαϊκής εποπτείας. Τι κάνει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση άμα δεν καταφέρνει να υπερασπιστεί τον Ευρωπαίο φορολογούμενο από απάτες τέτοιων διαστάσεων. Δηλαδή, μας παίρνουν τα λεφτά από τις τσέπες μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνει. Απλή και ξεκάθαρη ερώτηση. Μάλλον αυτή η ερώτηση θα έπρεπε να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές και όχι σε καθηγητές πανεπιστημίου και δημοσιογράφου, αλλά αν θέλετε να απαντήσετε μπορείτε. Έχουμε να κάνουμε με απάτη, με εγκληματικές ενέργειες και έχουμε παρατηρήσει ότι οι μηχανισμοί ελέγχου στα κράτη-μέλη και μεταξύ των κρατών μελών δεν υπάρχουν ή δεν λειτουργούν. Στην ε, ψηφιακή εποχή υπάρχουν στοιχεία για την κάθε μία ε, συναλλαγή με μετοχές και έχουμε παρατηρήσει ότι τέτοιες συναλλαγές έγιναν σε πολλές χώρες. Η Μεγάλη Βρετανία ήταν ε, στο επίκεντρο και φανταστείτε τι θα γίνει μετά το Brexit. Πρέπει να ακολουθήσουμε τα δεδομένα, πρέπει να ακολουθήσουμε τα, τα στοιχεία των ε, συναλλαγών διότι αυτές οι συναλλαγές είναι δυνατόν να γίνουν μόνο μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή όταν κατανέμονται τα μερίσματα. Και αυτό που είδαμε ε, και πάλι αναφέρομαι μόνο στην ε, πατρίδα μου, στην Γερμανία, είναι ότι δεν υπάρχει κανένας ελεκτικός μηχανισμός για, ε, την, για να ελέγξει τις, την καταβολή μερισμάτων. Και νομίζω πως θα έπρεπε να δημιουργηθεί ε, κα, κάποιος ε, μηχανισμός από πολιτικούς, από ε, ειδικού, έτσι ώστε να κλείσουν όλα αυτά τα παραθυράκια. Θα μπορούσα να προσθέσω κι εγώ κάτι ίσως. Α, συγγνώμη, δεν έχουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Και η ερώτηση ήταν πολύ μεγάλη, λυπάμαι, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο. ΕΛΚ, Σοσιαλδημοκράτες, ΕΛΚ, τώρα παίρνει το λόγο τα υπόλοιπα μέλη. Θα ξεκινήσουμε από το ΕΛΚ. Θα προτιμούσα να συνδυαστούν οι ερωτήσεις σας, αν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και θέλω να ευχαριστήσω και τους προσκεκλημένους μας ομιλητές. Θέλω να ε, τοποθετηθώ για αυτό που μόλις είπατε. Είπατε ότι υπάρχουν συστήματα ή ε, ελεγκτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι όμως ε, δεν έχουν επαρκείς αρμοδιότητες. Όπω η κατάσταση έχει διαμορφωθεί σήμερα πια, φαίνεται ότι οι φορολογικέ αρχέ μα δεν έχουν ούτε τι δυνατότητε ούτε τι αρμοδιότητε να μπορούν να παρεμβαίνουν γρήγορα και έγκαιρα λόγω των ραγδαίων τεχνολογικών ε, εξελίξεων. Ο κ. Μοσκοβισή έχει άλλωστε δηλώσει ότι ε, υπάρχουν ήδη μηχανισμοί και συστήματα για την ανταλλαγή πληροφοριών στα φορολογικά θέματα, αλλά δεν υπάρχει προθυμία να αξιοποιούνται από τα κράτη-μέλη αυτά τα συστήματα, αυτοί οι μηχανισμοί. Βεβαίως, πολλά κράτη-μέλη πλέον ε, ζητούν ε, τη διεύρυνση της ε, ανταλλαγής πληροφοριών στα φορολογικά θέματα για τη φορολόγηση μερισμάτων, την φορολόγηση κερδών από κινητές αξίες, δηλαδή και άλλους φόρους που υπερβαίνουν τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων. Θεωρείτε ότι αυτό θα ήταν μια χρήσιμη κίνηση, δηλαδή μια τέτοια διεύρυνση, ή θεωρείτε ότι υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. Δεύτερο ερώτημα. Πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες είχαν στο παρελθόν σοβαρά προβλήματα, όπως η Σανταντέρ, ερωτημα πολλες ευρωπαικες τράπεζε. ειχαν γιατί συμμετείχαν σε αυτού του είδους συναλλαγές της Κουμέξ. Όμως Πώ ωφελούνται από τη συμμετοχή του σε αυτές τις δραστηριότητε οι τράπεζες θεματοφύλακες. Ε, εισπράττουν κάποιες ε, ε, προμήθειε για την διενέργεια αυτών των συναλλαγών. πώ ωφελούνται. Πώς έγινε δυνατό η τραπεζική υποπτία να μην τσίμπησε τέτοιου είδου συναλλαγέ. Να μην τι εντόπισε για να τι ε, εμποδίσει. Και πώ θα μπορούσαμε να τι δώσουμε τι αρμοδιότητε για το μέλλον. Και τέλο. Είπατε ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο. Θεωρείτε ότι κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να συμβεί στη ΣΥΠΑ και στην Ιαπωνία, αν ναι γιατί, αν όχι επίση γιατί. Ποιος θέλει να απαντήσει. Ε, δεν, το, δεν το ξεκαθάρισα. Ο Τόμ έχει δύο σλότ, οπότε ε, τις συγχώνευσα. Ε, ευχαριστώ για την ανταλλαγή πληροφοριών πρώτα. Βεβαίω βεβαίως, ευχής έργων θα ήταν να υπάρχει ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών. Εμείς, για παράδειγμα, ως δημοσιογράφοι δημιουργήσαμε ένα διεθνές δίκτυο που ήταν πολύ χρήσιμο, ακριβώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών. Το γεγονός δε ότι ανάμεσα στη Γερμανία και στη Δανία για πάρα πολλά χρόνια δεν γινόταν ανταλλαγή πληροφοριών, ε, δείχνει ανάγλυφα ε, ποιο ακριβώς ήταν το πρόβλημα. Η δανέζικη κυβέρνηση, παρά το γεγονό ότι απίφθινε ερωτήματα στις ε, γερμανικές αρχές για πάρα πολλά χρόνια, δεν λάβανε απάντηση. Και επειδή και το φορολογικό απόρριτο στη Γερμανία είναι πάρα πολύ αυστηρό, ε, βεβαίω δημιουργούνται πάρα πολλά εμπόδια σε αυτή την ανταλλαγή πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση, ε, εγώ θεωρώ ότι η ανταλλαγή πληροφοριών πραγματικά πρέπει να διευρυνθεί ε, πέραν των, ε, του φόρου εισοδήματο φυσικών προσώπων και να περιλαμβάνει και τέτοιου είδου συναλλαγέ και τέτοιου είδου κέρδη. να προσθέσω κι εγώ κάτι. Εγώ θα πρότεινα να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών και μεταξύ των φορολογικών διοκτικών αρχών. Ή, εν πάση περιπτώσει, να συζητηθεί αυτό το θέμα. Γιατί σε πάρα πολλέ περιπτώσει βλέπουμε ότι οι επιτιθέμενοι είναι τα ίδια άτομα, οι ίδιοι κύκλοι. Για τη συμμετοχή των τραπεζών σε αυτές τις συναλλαγές, ως θεματοφύλακα, τράπεζα θεματοφύλακα. τίποτα δεν αποκομίζει ε, μια τέτοια τράπεζα. Όταν έχει τέτοιες ε, μετοχές στα χέρια της. Το μόνο πρόβλημα που δημιουργείται είναι ότι ευθύνονται οι τράπεζες αυτές για ψευδείς φορολογικές ενημερότητες και πιστοποιητικά. Ωστόσο, ο ρόλος, έχει δύο, ε, ο ρόλος των τραπεζών ε, έχει δύο όψεις αν θέλετε. Αφενός γίνονταν συναλλαγές με τις ίδιες τις μετοχές τους, με τα πακέτα των μετοχών των τραπεζών και δεύτερον από τις δικαστικές αποφάσεις που ελήφθησαν στη Γερμανία ε, αποδεικνύεται ότι οι τράπεζες αποφελήθηκαν από τη χρηματοδότηση τέτοιων συναλλαγών. Δεν ζητούσαν τόκο, αλλά ε, μερίδιο από τα κέρδη για την πραγματοποίηση και τη διευκόλυνση αυτών των ε, δραστηριοτήτων. ε, συμπληρωματικά να πω και εγώ ότι στις 18 ε, Οκτωβρίου η Γαλλία και η Ισπανία μάθαν από εμάς τους δημοσιογράφους ότι ήταν θύματα αυτών των συναλλαγών Κουμέξ ή Κουμκούμ. Και εμείς μόνο τα Κουμέξ files έχουμε στα χέρια μας. Δηλαδή τα ίδια έγγραφα που έχουν και οι φορολογικές αρχές. Ε, αναρωτιέται κανείς γιατί δεν έγινε ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, Γιατί δεν προειδοποιήθηκαν οι φορολογικέ αρχέ των κρατών μελών από τι ομόλογε του ε, αρχέ που τα μάθαν και τελικά χρειάστηκε να, έρθουν, να έρθουμε εμεί οι δημοσιογράφοι και να ενημερώσουμε τις, ε, τη Γαλλία και την Ισπανία. Ε, ρωτήσατε αν είναι κλασικό ευρωπαϊκό αυτό το πρόβλημα. Όχι, δεν είναι. Έχουμε δει και στην Ιαπωνία και στον Καναδά και στην, στην Νότια Αφρική τέτοιε δραστηριότητε δεν οροδούν προϋπήρων αυτές οι συναλλαγές. Ε, κάτι που βεβαίω δεν κάνει τα πράγματα καλύτερα, αλλά αξίζει να το έχουμε και αυτό κατά νου. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο και πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ, Υπερβάν Περέζ. Ευχαριστώ. Όταν λέτε ότι χρειάστηκαν 10 χρόνια για να συμπληρωθούν κάποια κενά σε μια χώρα που έχει ιδιαίτερα προηγμένη διοικητική ε, ικανότητα, αυτό μας ανησυχεί. Είπατε καταρχάς ότι έπρεπε να υπάρξουν ανταλλαγές πληροφοριών. Δεν ήταν μια μικρή θηκατρική, γιατί και πολλές, δύο φορές ο Ευρωπαίος Επόπτης προσπάθησε να βελτιώσει το σύστημα. Αλλά κατ' ουσία πώς εξηγείται ότι μια φορολογική αρχή και μάλιστα γερμανική και οι Δανέζικοι δεν ειδοποίησαν τις άλλες φορολογικές ε, αρχές απέναντι σε αυτό το κίνδυνο που είχε εντοπιστεί σαφώς και που ε, ε, είδαμε πως ήταν διασυνοριακός, κατεξοχήν διασυνοριακός. Και δημοσιογράφοι συνάδελφοί σας που συνέβαλαν στην έρευνα απαντούσε η φορολογική αρχή πολύ άσχημα ακόμα και όταν ε, τους ζητούσαν πληροφορίες άλλες φορολογικές αρχές. Πώς το αιτιολογείτε αυτό και έπειτα είδαμε στη Γαλλία το η Γερουσία ασχολείται με αυτό το θέμα και έχει ε, μάλιστα συσταθεί και στο Κοινοβούλιο μια ερευνητική επιτροπή ε, Άμεσα όμως έχει κατατεθεί και μια τροπολογία στο σχέδιο για τα ε, ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και λέει ότι τα έσοδα που προκύπτουν από την πούληση ενός μερίσματος σε έναν ε, αλλοδαπό δεν θα μπορεί ε, να δοθεί εκεί επιστροφή φόρων παρά μόνο εάν αυτός μπορεί να αποδείξει ότι είναι πραγματικός κάτοχος αυτού του μερίσματος. Προς τα εκεί κατευθύνεστε κι εσείς. Πιστεύετε πως μπορεί κάτι τέτοιο να επιτευχθεί και να τα καταφέρουμε χωρίς να έχουμε ένα εναρμονισμένο τέτοιο σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αν όντως χρειάζεται κάτι τέτοιο ποιο θα ήταν το κατάλληλο ευρωπαϊκό μέσο που θα έπρεπε να κινητοποιήσουμε. Έχω ακόμα μια ερώτηση, επιτρέψτε μου λίγο χρόνο ακόμα. Λέτε ότι οι τράπεζες αποθετηρίου όταν δεν ωφελήθηκαν αναγκαστικά, δεν κέρδισαν από αυτή την ιστορία. Αυτές οι τράπεζες, ε, ωστόσο, ε, εποπτεύονται ε, με πολύ ειδικό και ενισχυμένο τρόπο. Καμία όμως εποπτική αρχή δεν μπόρεσε να εντοπίσει αυτές τις συναλλαγές που είναι αρκετά μαζικές από ό,τι καταλαβαίνω. Ε, πώς έγινε αυτό, πώς οι αρχές δεν είδαν τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος θα ήθελε να ξεκινήσει. Η ερώτησή σας ε, είναι απόλυτα δικαιολογημένη, όπως και όλες οι ερωτήσεις ε, σήμερα. Ούτε και εγώ καταλαβαίνω γιατί χρειάστηκε τόσο πολύ καιρός έτσι ώστε να κατανοήσουμε τις συναλλαγές κουμέξ στην Γερμανία. Ούτε και καταλαβαίνω γιατί οι συναλλαγές κουμ-κουμ ε, συνεχίζονται ακόμα και τώρα στη Γερμανία. Επίσης, δεν καταλαβαίνω γιατί οι εποπτικές αρχές στη Γερμανία δεν ανέλαβαν την ε, εξέταση και τον έλεγχο των συναλλαγών αυτών. Ούτε και καταλαβαίνω γιατί την ε, περασμένη μόλις εβδομάδα έγινε γνωστό ότι μέσω πλαστών εγγράφων ε, υπάρχει ακόμα αυτή η επιστροφή παρακρατηθέντος ε, φόρου που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν υπάρχει αυτός ο ελεκτικός μηχανισμός και ε, δεν υπάρχουν μέτρα για να αποφύγουμε την ε, φορολογική απάτη. Το μόνο που θα μπορούσα να πω ως απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει ε, πολιτικό ενδιαφέρον για κάποια δυνατότητα να ληφθούν μέτρα μετά από συνεργασία. Συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να δούμε πού γίνεται παρακράτηση ε, φόρου εισοδήματος κινητών αξιών, ε, πώς ε, αποζημιώνονται, πώς, πότε επιστρέφεται πόσους, σε πόσες φορές. Νομίζω πως όταν κοιτάζουμε τα στοιχεία και βλέπουμε ότι κάποιος ε, έχει, ε, υπάρχει ανισορροπία στα έσοδα και έξοδα, τότε εντάξει δεν χρειάζεται και το φορολογικό σύστημα, το καταργήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Η Άννα Γκόμες έχει το λόγο. Έγινε και μια άλλη ερώτηση για την ε, πρόταση της Γαλλίας, για τη λύση που συζητείται αυτή τη στιγμή. Αν πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει κάποια λύση για να, μην, για να παρακρατάτε σε 30% για τους αλλοδαπούς ε, μετόχους, ο οποίος να επιστρέφεται μόνο αν ο μέτοχος αποδεικνύει με στοιχεία ότι είναι ο κύριος δικαιούχος της ε, μετοχής. Ακριβώς ε, αυτό. Αυτή είναι μια καλή αφετηρία. Να δούμε υπό ποιε προϋποθέσεις μειώνεται ένας φόρο, επιστρέφεται ένας φόρο και εκείνος ο οποίος υποβάλλει το, ερω... το αίτημα να του επιστραφεί η φόρος ε, θα πρέπει να αποδείξει με αξιόπιστα στοιχεία ότι το δικαιούται. Ακριβώς ε, αυτή είναι η μέθοδος, η λύση, η αρχή. Διαφορετικά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Η Άννα Γκόμες, τελευταία ομιλήτρια. Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σικ. Αν μπορεί να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Αν ακόμα εδώ. Α, όχι. Α, κάποιον άλλον τότε. Αν μπορούσε λοιπόν να επεκταθεί περισσότερο σε σχέση με το ρόλο της εποπτείας εθνικής και ευρωπαϊκής. Αν θα μπορούσε να είναι σημαντικός για να σταματήσει αυτό το σύστημα. Και ε, άλλη ερώτηση. Αν η Γερμανία απαγορεύει αυτό το σύστημα, το, απαγόρεψε το σύστημα το 2011, γιατί δεν ενημέρωσε τους υπόλοιπους. Τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, γιατί δεν ειδοποίησε τις εποπτικές αρχές σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο σε χώρες όπως η δική μου, όπου για παράδειγμα με, λόγω της Τρόικα έχουμε και αμνηστία ε, φορολογική του 2012 και έχουμε και ένα blackout φορολογικό ανάμεσα στο 2011 και το 2015 δηλαδή όλοι μπορούσαν να μεταφέρουν offshore χωρίς οποιοδήποτε έλεγχο στη διάρκεια της ε, ε, επιβολής της Τρόικα άρα οτιδήποτε μπορεί να έχει συμβεί εκείνα τα χρόνια για το ρόλο των εποπτικών αρχών. Από γερμανική εμπειρία να σας πω το εξής. Μέσα από τις έρευνές μας καταλήξαμε στο ότι η εποπτική αρχή ε, κεφαλαίου αγοράς ε, της Γερμανίας γνώριζε πάρα πολύ καλά ε, ποιοι είναι οι μηχανισμοί ε, που βρίσκονται σε εξέλιξη. Διότι ε, έπρεπε να εγκρίνονται, να, λαμβάνουν, να, να εγγράφονται στο, στο μητρό ε, φορολογικών ε, δραστηριοποιούμενων αυτές οι, αυτές οι, αυτές, αυτοί οι φορείς. Οι εποπτικές αρχές γνώριζαν, αλλά θεωρούν ότι δεν είναι αρμόδιες για φορολογικά ζητήματα. Κατά συνέπεια, οι προφορές αυτές δεν, κα, δεν κατέληγαν ποτέ στους αρμόδιους ε, της γερμανικής κυβέρνησης. Υπάρχει μια διάκριση δηλαδή ανάμεσα στις εποπτικές αρχές της κεφαλαίου και στις αρχές της φορολογικές. Δεν έγινε ε, εσωτερική ανταλλαγή ε, πληροφοριών. Και αυτό ήταν το λάθο και σε επίπεδο Γερμανία και βεβαίω και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί δεν μεταφέρθηκαν, δεν διαβιβάστηκαν αυτέ οι πληροφορίε. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Το, το κεφάλι μου μπορώ να κουνήσω μόνο. Υπόθηκε ότι και Γαλλία και Ισπανία ήταν ε, θύματα αυτών των συναλλαγών. Αυτό προκύπτει από τα αρχεία που έχουμε εμείς στα χέρια μας. Ε, για να τα έχουμε εμείς ε, στα χέρια μας αυτά τα αρχεία, μπορώ να φανταστώ ότι τα έχουν και διάφορες αρμόδιες αρχές. Επίσης, υπήρξε δικαστικό ερώτημα της Γερμανικής Εισαγγελίας προς την Ισπανία, που συνοδευόταν από επαρκή στοιχεία για το ότι η τράπεζα Σανταντέρ ε, διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο σε αυτές τις συναλλαγές και εκεί υπήρχε και η παράκληση ε, από τις γερμανικές αρχές να διερευνηθεί το θέμα. Υπήρχαν λοιπόν ε, επαρκή στοιχεία. Τι έκαναν οι ισπανικές αρχές. Διαβίβασαν το ερώτημα αυτό στην ίδια τη Σανταντέρ και τις ανέθεσαν εκείνης να απαντήσει στις γερμανικές αρχές. Πολλές φορές δηλαδή δεν μιλάμε απλά για ανεπαρκή ανταλλαγή πληροφοριών. Υπάρχουν και αρχές οι οποίες δεν ήθελαν την καυτή πατάτα στα χέρια τους. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω θερμότητα, θερμότατα τους ομιλητές μας, τον κύριο Σίκ που μας μίλησε μέσω βιντεοδιάσκεψης από το Bundestag, τον κύριο Σρόμ, τον κύριο Σαλέσκι, τον κύριο Σπέγγελ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και για την τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας δώσατε. Νομίζω ότι το βασικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε δυστυχώς είναι ότι όλα όσα μπορούσαν να αγνοηθούν δυστυχώς αγνοήθηκαν υπήρξε σοβαρή αμέλεια, είναι πραγματικά απίστευτη και όπως και σε τόσα άλλα ζητήματα η λύση είναι και εδώ στην ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών και καλύτερη συνεργασία μεταξύ χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Είναι ε, πολύ ενδιαφέρον. Πώς μπορούμε να χάσουμε τόσα πολλά πολύ δημόσιο χρήμα. Στις διαπραγματεύσεις ε, με το Συμβούλιο έχουμε την εντάξει οδηγία για τη διοικητική συνεργασία. Φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον για την εισαγωγή όλο ένα και περισσότερων στοιχείων που θα πρέπει να ε, ανταλλάσσονται. Ε, για να κλείσουμε νομίζω πως είναι ακόμα μια απόδειξη ότι που μπορούμε να δούμε ότι το φορολογικό μας σύστημα είναι πεπαλαιωμένο και δεν ε, είναι φτιαγμένο για τον 21ο αιώνα, ακόμα και για απλά θέματα και είναι καιρός να βρούμε καλύτερες λύσεις οι λύσεις δηλαδή που θα εξαρτώνται λιγότερο στη χώρα ε, από την κάθε χώρα, αλλά θα λαμβάνουν υπόψη μια ευρύτερη εικόνα. Εν πάση περιπτώσει, πέρασε η ώρα. Ευχαριστώ που κρατήσατε την πειθαρχία και τελειώνουμε στην ώρα μας. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες, τους ομιλητές ε, και θα τα πούμε στην επόμενη συνεδρίαση της ΤΑΚΣ 3. Καλό σας βράδυ